Buenas tardes. Lo primero, Καλησπέρα σας. Καταρχάς, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν γίνεται τακτικά. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς πάντα που παρόν. Θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια. Έχουμε μια αντιπροσωπεία βουλευτών της ΑΣΕΑΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε διερμηνία έτσι, ωραία. Καλωσορίζω. Τα αγγλικά πού είναι, πού είναι τα αγγλικά. Δύο, δύο λέει πρόεδρος. Δύο. Το βρήκε στο δύο. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Όπως λέγαμε, με χαρά καλωσορίζω την αντιπροσωπεία βουλευτών ΑΣΕΑΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας ε, επισκέπτονται από τις 10 μέχρι τις 12 σήμερα. και ήδη συνάντησαν του συναδέλφου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χθε το απόγευμα και σήμερα το πρωί συναντήθηκα με τον κύριο Λαμπρινίδη. Όπω ξέρετε, είναι οι χώρε τη Νότιο-Ανατολική Ασία, η ΑΣΕΑΝ, δημιουργήθηκε το 1967 κατά διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ για λόγου ασφάλεια. Και από τότε βέβαια αναπτύχθηκε και οικονομικά. Η ΑΣΕΑΝ είναι μια οργάνωση διακυβερνητική με ένα ισχυρό δόγμα μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των μελών και στην κυριαρχία τους. Αποτελεί αναφασβήτητα ένα από τους πιο ποικίλου οργανισμούς όσον αφορά τα, τα πολιτικά συστήματα, πολιτισμούς, οικονομίες κλπ. οι χώρε Μελή, Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ κλπ. Αυτή η σημερινή ανταλλαγή απόψεων θα επικεντρωθεί κυρίω στην περιφερειακή διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότερο από συγκεκριμένε δηλαδή εσωτερικές υποθέσεις. Θα θυμάστε ότι τον Οκτώβρη συναντηθήκαμε με την διακυβερνητική ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΑΣΕΑΝ δηλαδή το επίσημο όργανο της οργάνωσης αυτής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδρύθηκε το 2013 με στόχο την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες με ΑΣΕΑΝ. Δεν είναι επίσημο όργανο, αλλά ένα ανεξάρτητο όργανο. Καλό θα ήταν το επενθυμίσουμε αυτό, που συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε από βουλευτές με στόχο την αποτροπή των διακρίσεων, την προωθήση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Τα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνουν μάλλον είναι πολλά αναγνωρισμένα μέλη των κοινοβουλίων των χωρών αυτών με αναγνωρισμένη πορεία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε στοιχεία λοιπόν στους φακέλους σας και θα σας προσφέρω σύντομα αυτούς που έχουμε μαζί μας σήμερα. Μαλαισία Τσίλα Σαντιάγο, πρόεδρος αυτής της ε, οργανώσης, μέλος της αντιπολίτευσης στην χώρα του. Πριν την εκλογή του στο Κοινοβούλιο εργάστηκε σε ΜΚΟ. Η κυρία Μουσοσουά από την Καμπότζη, αντιπρόεδρος της ΑΣΕΑΝ είναι στο κόμμα που αποδεχθήκαμε εδώ τον Ιούνιο στην υποεπιτροπή μας. Ο κύριος Κάση Πυρώνια από την Ταϊλάνδη, διπλωμάτης, πρώην υπουργό Εξωτερικών από το 8 μέχρι το 11, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Ταϊλάνδης και τώρα είναι μέλος της Αναθεωρητική Συνέλευσης. Κυρία Σαϊβάρης από την Ινδονησία, από το κόμμα 5 είπε. Ιδρυτικό μέλος μιας ΜΚΟ, επίσης, που ασχολείται με τα θέματα των γυναικών στη χώρα της. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα με τις ομιλίες. Σας παρακαλώ να τηρήσετε τους χρόνους και καθυστέρησα, λυπάμαι, στο συγγνώμη, αλλά γι' αυτό έχουμε λιγότερο χρόνο. Κύριε Σαντιάγο, έχετε 10 λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αγαπητοί συνάδελφοι από τις χώρες θα σα φέρνω το μήνυμα της ειρήνης και της αλληλεγγύης από την ΑΣΕΑΝ και την Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σας ευχαριστώ για τις ασοικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ και την Υποεπιτροπή που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για το θέμα της ε, δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις χώρες ε, ΑΣΕΑΝ. Έχουμε 15 χρόνια εμπειρία στον τομέα αυτό, στη δική μας περιοχή του κόσμου. Έχουμε διάφορες εμπορικές συμφωνίες με ομάδες χωρών και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα εστιάσω την προσοχή μου σε τρία ζητήματα και συνάδελφοι σε άλλα. Εγώ θα ασχοληθώ λοιπόν με αυτέ τι εμπορικές συμφωνίε και το πώς επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να γύρω διασυνοριακά ζητήματα, όλο ιδιαίτερω. και μετά ε, να μιλήσω για τη διελκυστίδα των υπερδυνάμεων και πώς επηρεάζει αυτό το κράτος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό. Ποιε εμπειρικέ συμφωνίε ε, ε, διαπραγματευόμαστε και υπογράφουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε επαφή με χώρε ΑΣΕΑΝ αυτή τη στιγμή για την υπογραφή διμερών ε, εμπορικών συμφωνιών. Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ινδονησία και το καθεξής. Πριν από λίγα χρόνια ήταν ανομάδες χωρών, Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΣΕΑΝ. Υπεγράφει μια συμφωνία η οποία κατέρευσε και τώρα ακολουθείται μια διμερή διαφορετική προσέγγιση. Τι φοβούμαι εγώ. Ε, παρότι είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες, πρέπει να ενθαρρύνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των λαών της περιοχής. Διανοητικά και πνευματικά δικαιώματα. Αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Η συμφωνία 12 ε, χωρών με το μεγαλύτερο παίκτη της ΕΠΑ έχει 30 κεφάλαια και αυτή η Διατλαντική Συμφωνία περιέχει άκρος αμφιλεγόμενα κεφάλαια σε σχέση με την υγεία, τις θέσεις εργασίας, τον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και τις ίδιες της κοινωνίας. Θα δώσω ένα παράδειγμα για τα φάρμακα, παραδείγματος χάρη και τα πνευματικά δικαιώματα και για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι περισσότερες χώρες μας έχουν προσπογράψει τη Συμφωνία TRIPS. 20 χρόνια προστασίας ε, για, ε, για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Όμως, με τη συμφωνία τώρα επιτρέπεται παράταση ε, παόριστο της ισχύως ε, της προστασίας του διπλώματος. Δηλαδή, αυτοί που χρειάζονται προστασία δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα για να ε, επιβιώσουν. Λόγω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτό συνεπάγεται μονοπόλιο για τις εταιρείε και δείχνουν μελέτες πόσο οι εταιρείε μπορούν να έχουν επιστροφή της επένδυσης σε 3-4 χρόνια. Τα υπόλοιπα είναι υπερκέρδη για τις εταιρείε. Μπορώ να σας δώσω πληροφορίες. Προκύπτει με σαφήνεια από αυτά τα στοιχεία ότι εκμεταλλεύονται τα μιανωτικά δικαιώματα για αυτά ε, τα υπερβολικά ε, κέρδη αντί να έχουν ε, πρόσβαση οι άνθρωποι που τα χρειάζονται, οι άρρωστοι που τα χρειάζονται χρειάζονται σε φάρμακα σε προσιτές τιμές, ε, κάτι που είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Στη Μαλαισία, ένα στους τέσσερις ε, μέχρι τα 35 θα πάθει καρκίνο. Ε, καρκίνο του μαστού, μία γυναίκα στις 40. Πώς ε, θα προστατευτούν με αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνία γιατί υπάρχει υπέρβαση της 20 για την προστασία των φαρμάκων βάσει αυτών των διατάξεων. Γι' αυτό θα ήθελα να εξετάσουμε και αυτή τη διάσταση της πρόσβασης στα φάρμακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Δεύτερον, διασυνοριακά ζητήματα, μετανάστευση, πρόσφυγες, εμπορία ανθρώπων και ε, ε, ε, την σύμβαση ε, την έχουν υπογράψει οι Καμπότζοι και οι Φιλιππίνες για τους πρόσφυγες. Νομίζω υπάρχει δυνατότητα ρύθμιση ώστε να υπογράψουν και να προσχωρήσουν και άλλες χώρες. Διότι στη Μαλαισία, παραδείγματος χάρη, ε, υπάρχει μεγάλη προσέλευση προσφύγων, δεν χαίρουν όμως καμίας προστασίας, μηδενικής προστασίας και εάν χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο, είναι υπερβολική η τιμολόγηση, δηλαδή αντιστοιχεί σε ε, μονόκλινο για, τον, ε, για το Μαλαισιανό, παραδείγματος χάρη τιμές. Ε, λοιπόν, ε, ρουχισμός, στέγη, τροφή, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Μετανάστευση. Είμαστε παράδεισος για τη μετανάστευση. Ε, τέσσερα εκατομμύρια μετανάστες εργάτες, στη Μαλαισία δύο εκατομμύρια. Και ε, εισάγουμε και εξάγουμε τέτοια, τέτοιες, ε, τέτοιους εργάτες μετανάστες. Ε, Χρειαζόμαστε την προστασία λοιπόν των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει μια σχετική δήλωση, έχει υπογραφεί μόνο από δύο χώρες και νομίζω θα πρέπει να το θέσουμε και αυτό το ζήτημα. Εμπορία ανθρώπων. Ε, υπάρχει δήλωση ε, επίσημα, αλλά είναι κενή ε, ουσίας. Δεν έχει αναλυθεί καμία δράση. Ε, θα παρακολουθήσατε τι έγινε στη Μιανμάρ ε, για τη βία κατά της ε, μειοψηφικής ε, πληθυσμιακής ομάδας. που αναγκάστηκε να αποχωρήσει ε, και στην Ταϊλάνδη και στην Ινδονησία θα μπορέσουν τελικά να βρουν κάποια βοσκοτόπια για να επιβιώσουν. Ε, αναγκάζονται να αποχωρήσουν και κατευθύνονται προς την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη. Αυτό ε, αυτή τη μετακίνηση την αναλαμβάνουν αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι όμως συνεργάζονται με κυβερνητικούς ε, οργανισμούς ε, που υποτίθεται προστατεύουν τα συμφέροντα του κράτους, αλλά τελικά αυτές οι αρχές συνεργάζονται με τους διακινητές. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό. Είναι κοινή γνώση στις χώρες μας ότι οι αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται με τους διακινητές. Υπάρχουν δημοσιεύματα που δείχνουν ότι 80% των υπαλλήλων ε, εμπλέκονται σε δύο υποθέσεις συνεργασίας με τους διακινητές ε, ούτως ώστε ε, γυναικόπαιδα και άντρες να μπαίνουν στην Μαλαισία. Μία νέα γυναίκα 23 χρονών επιβίωσε από την Πόκο Χαράμ και μετά πήγε στη Μαλαισία και λόγω των διακινητών έχει πέσει θέμα της βιομηχανίας του σεξ στη Μαλαισία και είναι ζει σε συνθήκες δουλείας. Υπάρχουν ε, πρωτόκολλε συμφωνίες ε, που χωρίς κανένα πρόβλημα υπογράφει η κυβέρνηση, αλλά σε, στον τομέα της επιβολής μηδέν, είναι τα αποτελέσματα. Ε, ε, θρησκευτικός εξτρεμισμός τώρα. Υπάρχουν πολλά είδη. Μιλάμε για τον φονταμεταλισμό του Ισλάμ. Όμως στην Ανατολική Ασία έχουμε και βουδιστές φονταμεταλιστές ε, που είναι πάρα πολύ βίαιοι στη Μιανμάρ παραδείγματο χάρη ε, το πώς μεταχειρίζονται τους Ροχάνους παραδείγματος χάρη αυτή τη μειοψηφία στο, στο Μιανμάρ. Και στην Τελάνδη αλλά και στη Σρι Λάγκα ε, συνεργάζονται με συντηρητικέ αντιδραστικέ ε, δυνάμει ε, για να ξεκινήσουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό με κηρύγματα μίσου. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται για παστικισμό. Ένας άλλος θρησκευτικό φονταμαντελισμός. Ε, ποια είναι η παγίδα. Οι άλλες κυβερνήσεις άλλο χωρών χρησιμοποιούν αυτόν τον εξτρεμισμό για να ποινικοποιήσουν ε, να ποινικοποιήσουν θεμητή εθνοτική προέλευση. Ε, ε, αυτό που ήθελα να πω είναι αυτή η διελκυνσίδα των υπερδυνάμεων στην περιοχή. Τρεις είναι, είπα από τη μία, Κίνα από την άλλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. έχουν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα την τελευταία διετία που μια υπερδύναμη σήμερα μπορεί να εξαγοράσει και τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για να εξυπηρετήσει την εξωτερική της πολιτική, τα οικονομικά ή γεωπολιτικά της συμφέροντα στην περιοχή. Οι υπερδυνάμεις Ε, μέσα από στρατιωτική οικονομική βοήθεια υποστήριξη για τις υποδομές ε, ε, επιβάλλουν τις επιταγές τους στις κυβερνήσεις και είναι και τόσο δημιουργικές που μπορούν να χρησιμοποιούν σαν χειρανθρώπους σε πολιτικές φυσιογνωμίες και να καθοδηγούν την πολιτική ζωή στις χώρες ΑΣΕΑΝ. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Υποτίθεται ότι είναι μια ζώνη ουδέτερη, μια ζώνη, μια περιοχή του κόσμου ειρηνική. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ουδετερότητα δυστυχώς ε, στις διπλωματικές σχέσεις των χωρών της ΑΣΕΑΝ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά υπερβήκατε το χρόνο σας, λέει η Πρόεδρος. Αχα, τότε θα συνοψίσω να πω πως κινδυνεύει η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες Ασιαν. Έχουμε φτάσει ε, στο σημείο μη επιστροφής και νομίζω ότι θα πρέπει να δράσουμε όχι μόνο προς συμφέρον των χωρών Ασιαν αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σας ευχαριστούμε. Μη σας ευχαριστούμε κύριε Σαντιάγκο. Μας τα είπατε αναλυτικά και περιγραφικά για τα καταλάβουμε. Ιδιαίτερα στους τομείς που αναφερθήκατε διεξοδικά. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους βουλευτές που είναι στην αίθουσα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πείτε μου αν θέλετε πάντως να μιλήσετε για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Η κυρία Λόκη Πιλέρ, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβα καλά. Θα ακούσουμε και από... Θα μιλήσουν και αυτοί που βρίσκονται στο πάνελ. Είναι μόνο ερωτήσεις στον πρώτο μιλητή. Μπορείτε να ρωτήσετε όλους τους ομιλητές. Θα δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους στο πάνελ. Ο κύριος Σαντιάγο μας έδωσε μια γενική προσέγγιση. Μπορείτε να ρωτήσετε που θα μπορέσουν μετά να απευθυνθούν και στους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστώ για την δήλωση, για την ανακοίνωση και για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής οργάνωσης. Ρωτήσατε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να υπογράψουν στην πρόσφαση ένα γράμμα για να αφαιθούν ελεύθεροι ε, κρατούμενοι συνείδηση. Και αυτό είναι κάτι που το καλωσορίζουμε ως πρωτοβουλίο. Όσοι δεν έχουν υπογράψει ας το κάνουν, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό. Κύριε Σαντιάγο, είπατε ότι αποτύχατε να έχετε μια κοινή διακήρυξη για την προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους. Θα μπορούσατε λίγο να το εξηγήσετε αυτό λίγο περισσότερο. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ε, για τις οικογένειες των μεταναστών. Υπάρχει μια διστακτικότητα εδώ και 15 χρόνια. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η δική σας εμπειρία όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί φέτος την πολιτική ενάντια στο τράφικινγκ εντός και εκτός της Ένωσης. Μπορούμε να σας δώσουμε μια έκθεση πριν το καλοκαίρι για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πιο εντατικά για να καταπολεμήσει ε, την εμπορία ανθρώπων στο εξωτερικό της. Πρέπει να ακολουθήσουμε και την πορεία των χρημάτων ε, αυτής της δραστηριότητας, τα οποία καταλήγουν σε ευρωπαϊκές τράπεζες. και στα διάφορα ψηφίσματά μας απ' έξω φαίνεται ότι όλη η περιοχή έχει ένα πρόβλημα με την θανατική ε, καταδίκη. Είναι κάτι που προκύπτει πολύ συχνά. Πρόσφατα υφετήσαμε ένα ψήφισμα για τις Φιλιππίνες σε σχέση με αυτό το θέμα και θα ήθελα να ακούσω και από εσάς πώς αντιμετωπίζει το δικό σας ε, δίκτυο ε, το θέμα της θανατικής ποινής. και πώς θα οδηγηθούμε στην κατάργηση. Και μετά έχουμε τα θέματα της ε, αφαίρεσης ε, ιδιοκτησίας γης. Υπάρχει ένα ψήφισμα και γι' αυτό, την κατάσχεση μάλλον ιδιοκτησίας. Από το 2003 πάνω από 4.000 ε, ε, κάτοικοι της υπαίθρου έχουν ε, θυχτεί από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η αρπαγή της γης και η έλλειψη σχετικής νομοθεσίας σε πολλές χώρες είναι και αυτά θέματα που θα πρέπει να σας απασχολήσουν. Πριν από δύο εβδομάδες, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια οργάνωση για την προστασία εξέθεσε, έκανε μια έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο για α, δολοφονίες στην Ταϊλάνδη που σχετίζονται και με θέματα ιδιοκτησία γης. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα που συρρυκνώνεται ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών. και ο εκπρόσωπο τη ε, Ταϊλάνδη και τη Ινδονησία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μα μιλήσει γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πετίνη. Έχετε το λόγο. Σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς τους βουλευτές που μας επισκέπτονται. Μιλήσαμε στην αρχή για την ποιότητα της δημοκρατίας της χώρας ΑΣΕΑΝ. που είναι ισχνή και υπάρχει κίνδυνος επιστροφή στο παρελθόν. Τι άποψη έχουν όμως οι προσκεκλημένοι μας για την κατάσταση στη Βυρμανία και τη δημοκρατία εκεί. Τι άποψη έχουν επίσης για την έγκριση του νέου συντάγματος της Ταϊλάνδης που πέρασε από διάφορα στάδια, από 40 κύματα. Αλλά τουλάχιστον τώρα φτάσαμε σε κάποια ανηνεμία, τουλάχιστον βλέποντας το απ' έξω. Και τέλος, τι έποψη έχουν για τον νέο πρόεδρο των Φιλιππίνων. Γιατί έχουμε κάποιες μαρτυρίες στην Ευρώπη ανησυχητικές. Θέλετε κάποιος λοιπόν να εμβαθύνετε για αυτά τα ζητήματα και που δείχνουν ότι τελικά δέχεται πίεση τη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Μια και δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο, να κάνω και εγώ δύο σύντομες ερωτήσει στους προσκεκλημένους μας. Ηρώνια πρώτα, από την Τελάνδη. τι θετικό μπορούμε να περιμένουμε από την βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών που θα έχουμε και την Ιαία Μογκερίνη αυτή τη βδομάδα για τον κύριο Μπέρενς. Λόγω της εμπειρίας σας για τα θέματα ισότητας και σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Σαντιάγο για τα πνευματικά δικαιώματα και την πρόσβαση ας πούμε στα φάρμακα. και τα μονοπόλια που υπάρχουν. Ποιες κοινέ δράσεις θα μπορούσαμε να ευθετήσουμε για να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση ανδρών και γυναικών, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ούτε καν στις ε, κλινικές δοκιμές δεν υπάρχει αυτή η ισότητα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε από κοινού εμείς και εσείς για να βελτιώσουμε αυτό το μοντέλο. Για να βελτιώσουμε δηλαδή όχι μόνο τη διαφάνεια αλλά και την επαναφορά, την επιστροφή των κονδυλίων στην έρευνα. Θα σας δώσω τώρα το λόγο να απαντήσετε δύο λεπτά ο καθένας. Στο συγγνώμη για το σύντομο τις ομιλίες σας, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εσά. Ο κ. Σουκώ έχει το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για την υφαρπαγή γεών στην Καμπότζη όχι μόνο στην περιοχή ΑΣΕΑΝ είναι μείζον ζήτημα. Ε, η φαρπαγή γιών στα πλαίσια της ανάπτυξης και το πώς γίνεται ακριβώς. Στην ε, Καμπότζη είναι μέσα από την πολιτική των εκχωρήσεων γεών. Παίρνουν γη από τους μικρούς γεωργούς, ώστε παράνομα να τη δώσουν στις μεγάλες εταιρείες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά Κάποιες εταιρείε παράγουν προϊόντα όπως ε, ζάχαρη, παραδείγματος χάρη, που εξάγεται συνέχεια σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει τη συμφωνία ε, όλα εκτός από όπλα. Έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα, τους γεωργούς ε, που πέφτουν θύματα αυτών των εκχωρήσεων. πλήττονται στην καθημερινή του ζωή. Δεκάδες, χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια γεωργοί έχουν πληγεί. Είναι σοβαρότερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών. Επιτρέψτε μου εντάχει να μιλήσω και για τη Βυρμανία και να εξηγήσω πως κατήγαγε το NLD μεγάλη νίκη, η κυρία Άνσου Μεγάλη δύναμη των δημοκρατικών δυνάμεων. Στην Καμπότση και σε άλλες χώρες του ΑΣΕΑΝ υπάρχει δίψα για δικαιοσύνη, για δημοκρατία. Αυτό είναι υπαρκτό και ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε, να μας υποστηρίξετε, να σταθείτε στο πλευρό των ε, δημοκρατικών δυνάμεων, από πλευράς ε, των ε, μελών των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων των χωρών Ασιών. Σας ευχαριστούμε για το ψήφισμα για την Καμπότζη που εγκρίνατε στην Ολομέλεια. Ζητούμε δε επιβολή στοχευμένων κυρώσεων για τις θεωρήσεις, παραδείγματος χάρη. Και Ε, για να περάσουμε ένα μήνυμα στο δικτάτορα της Καμπότης και σε άλλους δικτάτορες ότι ε, δεν μπορούν ε, να περνάνε ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Πυρόμια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. ψήφισα ενάντια στο Σύνταγμα και το δημοψήφισμα που έγινε για την ειδική σύγκλιτο και είπα ναι δημοσίως στον τύπο στην ε, Εθνική Συνέλευση για τις Μεταρρυθμίσεις αλλά αλλά είναι μια ελεγχόμενη δημοκρατία με την παρουσία του στρατού στην Άνω Βουλή και στρατηγικό πρόγραμμα 20 ετών και ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει εκπονηθεί από το στρατό. Θεωρώ ότι ο κόσμος της Ταϊλάνδης, οι άνθρωποι της Ταϊλάνδης πολίτες και της υπόλοιπης Ασίας έχουν φιλοδοξίες να ζήσουν ε, σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον και πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμούμε γι' αυτό. Στον αγώνα αυτό ίσως δεν μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας. Ίσως χρειαζόμαστε βοήθεια. Θα πρέπει να μας βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε να στείλετε στρατό, αλλά μπορείτε να βοηθήσετε, να βοηθήσετε στην δημιουργία θεσμών, να ε, συνεχίσετε μαζί μας στην πολιτική και κοινωνική αγωγή έχοντας ως παράδειγμα την εκδημοκρατικοποίηση της Ανατολική Γερμανίας όταν ε, αποσχίστηκαν από την ε, Σοβιετική Ένωση, βγήκαν από την σφαίρα επιρροής. και να ενισχυθούν οι δημοκρατίες σε όλες τις χώρες της Ασίας. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η φύση των μελλοντικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ταϊλάνδης. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση ανάμεσα στον, στην στρατηγική κυβέρνηση και τη σχέση με τον λαό σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διαπραγματεύσεις για, για την ε, Συμφωνία Ελευθεροπορία, η οποία αναστάλθη λόγω του στρατού. Στείλαμε ένα σημείο σημείωμα στον ε, Επίτροπό σας να συνεχιστεί η τεχνική διαβούλευση αλλά για να συνάψουμε συμφωνία ελευθέρω μπορεί θα πρέπει να γίνει με μια δημοκρατική κυβέρνηση και όχι μια στρατική κυβέρνηση. Θα υπεγραφεί το θα έχουμε ένα πλήρως δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα. Θα... Η πρόεδρος παρακαλεί τον ομιλητή να ολοκληρώσει. το. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπαρέντς. Δύο ερωτήματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο σχετίζεται με την φαρπαγή γεών στην Ινδονησία. Είχαμε τέτοια περιστατικά πρόσφατα. Με βάση τη διεθνείς Συμφωνία Επενδύσεων, η κυβέρνηση της Ινδονησίας Έχει 18 διμερείς ε, συμφωνίες. για να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ε, προστασία των επενδυτών και την εθνική κυριαρχία. Οι διατάξει των περισσότερων ε, συμφωνιών, συμφωνιών είναι απαρχιωμένες γιατί δεν ε, αφήνουν πολύ μεγάλο περιθώριο στις χώρες ε, για να ξέρουν πώς θα ε, διεξαχθούν όλα αυτά τα προγράμματα επενδύσεων. right national ναι, και το πρόβλημα είναι το σύστημα ESDS μέσα στις εμπορικές συμφωνίες για την προστασία των παιδιών και τις σχέσεις τους με τις κυβερνήσει των κρατών μελών. Ε, και γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή σα σε αυτέ τι διατάξει συμφωνίε, γιατί επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων κυρίω για τα πολιτιστικά του δικαιώματα γιατί θεωρούμε ότι ε, ε, περί αυτού πρόκειται να μιλάμε για το δικαίωμα στη γη. Τώρα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα σε σχέση με την μεταρρύθμιση και την ε, ανακατανομή ε, των γεωτεμαχίων ε, για τον τόπιο πληθυσμό, τον αυτόχθονο πληθυσμό και σχετίζεται με την επιζητιστική ασφάλεια. Είναι καλό αυτό το πρόγραμμα για μας, διότι... Μεγάλο κομμάτι της γης, πώς το λένε, Ε, ε, έχει η ε, φαρπαγή από μεγάλες επενδυτικές εταιρείες στην Ινδονησία. Το δεύτερο πρόβλημα που μας απασχολεί στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία στο Κοινοβούλιο είναι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή ε, στην κατοχήρωση των ατομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων έχουμε ισχυρό νόμο προστασίας των ε, δικαιωμάτων των γυναικών κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ε, της σεξουαλικής βίας, αυτό προετοιμάζουμε τώρα. Νομίζω να σταματήσω εδώ γιατί μου λέει ότι δεν έχω χρόνο. συγγνώμη λευρός που σας πιέζω. αλλά μην ανησυχείτε, όλοι λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που μας δώσατε. Κύριε Σαντιάγκο, δύο λεπτά έχετε για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στα ερωτήματά σας ε, για την πρόσβαση στα φάρμακα. Ε, στον ε, ακαδημαϊκό χώρο αλλά ε, και στις, ε, στους ασθενείς ε, και στις ομάδες ασθενών Αναπτύσσεται αυτή η τάση υπέρ του αξιώματος ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αγαθό η πρόσβαση στα φάρμακα. Johnson και Τζόνσον, παραδείγματος χάρη. 8,2 δις δαπάνης από το 2014 για την έρευνα. 17,5 δισεκατομμύρια για τις ε, πωλήσει και το μάρκετινγκ. Βλέπετε το χάσμα. 8,2 ε, για την έρευνα και τα διπλάσια για τις ε, πωλήσει και το μάρκετινγκ. 13,2 δις κέρδη. Κερδοσκοπία είναι αυτή, δηλαδή εις βάρος κυριολεκτικά της υγείας των ανθρώπων έχουν αυτά τα κέρδη. 22 δις ε, από την πώληση φαρμάκων. Νομίζω ότι... Ναι, είναι θεμητό να θέλουν επιστροφή των επενδύσεων, όμως δεν μπορεί να έχουν κέρδη 22, ύψους 22 δις. Και επειδή το θέσατε το ζήτημα, Ε, ο φόβος ε, έχει επικρατήσει στην περιοχή και σας το έλεγα και πριν, πενικοποιείται θεμητή εθνοτική προέλευση σε πολλές χώρες. Ε, στη Μαλαισία, ε, το 1 τρίτο θα μπει φυλακή εάν η κυβέρνηση τους διώξει μέσα αυτού του νόμου sedition προδοσίας όπως ονομάζεται Ε, υποτίθεται ότι αυτή η δημοκρατία και διαρκώς παράγονται νέα νομοθετήματα για να παραβιάζονται τα δικαιώματα κάποιων και να ελέγχουν τις κοινωνίες. Η... Πού είναι η βουλευτήνα Λόχμπιλερ, ήθελα να της πω ότι αυτή η δήλωση ε, της ΑΣΕΑΝ ναι, γιατί δεν εφαρμόζεται στη Μαλαισία μπορώ να σας πω τι γίνεται με, την μετανάστευση. Ο αριθμός των θανάτων ε, σε μετανάστες εργότες που κρατούνται είναι τόσο υψηλός ε, που τι να σας πω, ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και λένε κάποιοι τι, θέλουμε τη δήλωση τότε. Λένε λοιπόν άλλοι ότι είναι αδήλωτοι, δεν έχουν έγγραφα αυτοί οι εργάτες και υπολογίζει ο τους σε 2 με 3 εκατομμύρια. Εάν η Μαλαισία την υπογράψει αυτή τη συμφωνία, τότε ε, εμείς ευθυνόμαστε που ε, εξάγεται αυτό το εργατικό δυναμικό ε, αδήλωτα. Πώς γίνεται όμως να θα παραμείνουν στη Μαλαισία, δεν γίνεται αυτό, λόγω της διαφθοράς. Αυτή η διαφθορά τρώει σαν και όλο το κράτος, φτάνει μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης. και θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά, ώστε να επιτύχουμε έναν εκδημοκρατισμό στην ε, Μαλαισία, γιατί πραγματικά είμαστε σε δινή κατάσταση. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σε αυτό το πάνελ. Ήταν πολύ χρήσιμο που ακούσαμε την εμπειρία σας και τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Επικεντρωθήκατε μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο συγγνώμη για την πίεση, αλλά δυστυχώ αυτούς του ρυθμού έχουμε. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι χαιρόμαστε κάθε ευθερόλεπτο των ομιλίων σα. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Για την επόμενη συνεδρία και κλεισμένων παρακαλώ τους μη συμμετέχοντες να φύγουν ώστε να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατό.